Ο κύριος Έριξον ε, διορίστηκε στην ε, σουηδική κυβέρνηση και γι' αυτό λοιπόν το συγχαίρουμε. Και έτσι λοιπόν ε, από 25 Μαΐου χείρεψε